Colleagues, if I can bring the meeting to order, I know we're a little. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Έχουμε καθυστερήσει λίγο. Ήθελα να δώσω τη δυνατότητα στους συναδέλφους να έρθουν ε, στη συνεδρίαση, γιατί υπάρχουν και τα οδοφράγματα έξω. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη έχουμε την έκθεση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ε, την οποία θα μας κάνει η κυρία Ζακλίν Μαγκλέιτ, ε, παρουσίαση της έκθεσης τέρμου. Κυρία Μακλέιτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και πάλι εδώ στην Επιτροπή σας. Έχετε λοιπόν την έκθεση ΤΕΡΜ ενώπιόν σας. η οποία αναλογεί και στα όσα είχατε γράψει στο ψήφισμα για την ε, Λευκή Βίβλο των Μεταφορών ε, το 2011 που μας είπατε ότι θα πρέπει να ε, λάβουμε μέτρα για να επιτύχουμε τους στόχους και αυτό προσπαθεί να σας παρουσιάσει η έκθεση. Να σας πω το εξής. Το εξώφυλλο ε, προέκυψε μέσω διαγωνισμού ο οποίος έγινε και υπήρξε και δημόσια ψηφοφορία και ο νικητής είναι ένας ε, νεαρός Ισπανός, ο οποίος τράβηξε αυτή τη φωτογραφία και θα του δοθεί ένα βραβείο ε, με την παρουσία του Επιτρόπου Ποτότσνικ το Φεβρουάριο. Να περάσουμε όμως την έκθεση αυτή καθεαυτή. Το 2013, όπως γνωρίζετε, είναι το έτος ε, του αέρα. Γι' αυτό λοιπόν επικεντρωνόμαστε στις μεταφορές και τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα του αέρα και το πώς επιδρά αυτό στον ανθρώπινο πληθυσμό θα πρέπει να πούμε ότι οι μεταφορές εξακολουθούν να είναι υπεύθυνε για μεγάλα ποσοστά ρήπανσης και ε, αέρια εκπομπών, ε, ε, εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Επομένως, εξακολουθεί να αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα σε σημαντικούς τομείς. τα αυτοκίνητα οχήματα δεν έχουν επιτύχει να κάνουν πραγματική μείωση του διοξιδίου του άνθρωπου και αυτά τα επίπεδα μας ανησυχούν και στην νομοθεσία, αλλά υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στην ποιότητα του αέρα συνολικά. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια ως προς το τι ε, οδηγεί στη χαμηλή ποιότητα του αέρα είναι οι εναέριες μεταφορές και αυτό είναι και ε, ε, η αιτία των μεγάλων ποσοστών διοξιδίου του αζότου. Η όξινη βροχή επίσης μειώθηκε μόνο κατά 14% από το 1990 παρά τις μεγάλες ε, βελτιώσεις που έγιναν σε θέματα απόδοσης. 14% διορθώνει ο Μιλήτρια. Για τη συνολική εικόνα λοιπόν του 2012, 2010 ε, συγγνώμη, μπορούμε να δούμε κάποιες βελτιώσεις, αλλά ε, θα πρέπει να το δούμε στο σύνολο των αερίων του φαινομένου του θερμοκυπρίου, που είδαμε ότι είχαν μειωθεί το 2010, αυτό ε, το ε, αποδώσαμε στην ε, ύφεση και οι τιμές που βάλαμε το 2011 μας δείχνουν ότι έχουμε μια συνολική μικρή αύξηση στα αέρια φαινομένων του θερμοκηπίου. Και επομένως βλέπουμε ότι ναι μεν η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ε, συνεχίζονται κάποιες ε, πηγές ρήπανσης στις αέριες μεταφορές και θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα από αυτού. Η αύξηση ενέργειας για τις μεταφορές αύξησε, αυξήθηκε το 2011 σε σχέση με το 2010, αλλά οι εκπομπές ε, του 2010 μειώθηκαν μόνο κατά ένα μικρό ποσοστό, 0,5% σε σχέση το, με το 2009. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι είναι σταθερές αυτές οι εκπομπές. Τώρα, πολλοί από του άλλου στόχου δεν έχουν κινηθεί καθόλου προ τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε κάποιες βελτιώσεις ε, στις εκπομπές ε, από τα νέα αυτοκινητά οχήματα, επιβατηγά, αλλά δεν έχουμε μειώσει την ε, κατανάλωση των καυσίμων για τις μεταφορές και είχαμε και ένα στόχο 10% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν έχουμε επιτύχει και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Δυστυχώς ε, ε, για τα ηλεκτρικά οχήματα, παρά το γεγονός ότι στα ποσοστά φαίνεται καλό, τα αποτελέσματα είναι μάλλον μέτρια. Το 2002 είχαμε ένα αυτοκινητόχημα ηλεκτρικό, ε, όσον αφορά στις πωλήσει τώρα είμαστε στις 7.000 πωλήσει ηλεκτρικών οχημάτων το 2010 και το 2011 είχαμε 9.000 οχήματα. Τα ποσοστά λοιπόν φαίνονται καλά, στην πραγματικότητα όμως για τον στόλο που έχουμε στους αυτοκινητοδρόμους είναι πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό. Έχουμε κάποιε καινοτομίε στην τεχνολογία για τι μπαταρίε, διάφορε μορφέ κινητήρων και κ.ο.κ. Επομένω, σαφώ ε, αρχίζει να προβάλλει κάτι καλό, αλλά δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα ε, θα ενταχθούν όλα αυτά ώστε να έχουμε ένα στόλο ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τώρα, οι εκπομπέ φαινομένου θερμοκηπίου για τι μεταφορέ σε πραγματικού όρου, είναι ε, ένα 6% πάνω από τα επίπεδα, συγγνώμη, 26% πάνω από τα επίπεδα του 1990. Αυτό περιλαμβάνει και τις εναέριες μεταφορές και αυτό που βλέπετε από το διάγραμμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες σαφείς πτώσεις, πολύ χρήσιμες, αλλά αν δείτε ε, στην πάνω γραμμή έχουμε το διοξίδιο του θείου, το οποίο μειώνεται, μειώνονται τα αιωρούμενα σωματίδια, αλλά αν δείτε ε, τι γίνεται με το διοξίδιο του αζότου, τότε βλέπετε ότι είναι σημαντικό το, σωστό ε, το ποσοστό και θα έπρεπε να επικεντρωθούμε σε αυτό, διότι όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, το διοξίδιο του αζότου είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι έχουμε μειώσεις σε πόλεις και η έκθεση περιλαμβάνει και μία ανάλυση 40 πόλεων, επομένως έχουμε πολύ συγκεκριμένα σημεία στα οποία επικεντρωνόμαστε εδώ, ε, κοιτάμε τις αναλογίες από πόλεις και αν δούμε μία πόλη όπως για παράδειγμα η Γλασκόβη, διαπιστώνουμε ότι το διοξίδιο του αζότου εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Οι μεταφορές ε, βέβαια είναι η βασική αιτία και βλέπουμε ότι Κατά 44% υπερβήκαμε τους, τα ποσοστά για το διοξίδιο του αζότου. Και γιατί μας ανησυχεί αυτό, διότι είναι ο προπομπός του όζοντος, που είναι αυτό το οποίο επηρεάζει σημαντικά την ανθρώπινη υγεία. Στα αερούμενα σωματίδια 10, το PM10, το οποίο γνωρίζει το κοινό, έχουμε το 33% ε, άνω από το ποσοστού, αλλά ξέρουμε ότι αυτό έχει συνέπειες για το καρδιαγγειακό σύστημα και ούτω καθεξής. Σε γενικές γραμμές λοιπόν είμαστε ακόμα σε πολύ σημαντικά επίπεδα στις πόλεις και διαπιστώνουμε ότι οι μεταφορές αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και έχουμε έκθεση σε πολύ υψηλότερα ποσοστά από τις ε, ε, κανονικές τιμές. Να πω λίγα πράγματα για την αυσιπλοεία. Εδώ διαπιστώνουμε ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα εικόνα στην αριστερή πλευρά. Έχουμε όλες τις μεταφορές και στη δεξιά πλευρά έχουμε την αυσιπλοεία. Κρίμα που δεν έχουμε τους δρόμους του Ρόντερνταμ, αλλά βλέπετε εδώ πέρα ε, την πραγματικότητα, τη συγκέντρωση αιρούμενων σωματίδιων. Είναι πολύ σημαντικό ποσοστό, 9 και 12% σε σχέση με το 1997-2003, ε, αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντική πηγή ε, διοξιδίου του, του θείου που είναι 19% των εκπομπών του 2010. Η ναυσιπλοεία λοιπόν εξακολουθεί να μας απασχολεί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες μειώσεις ε, λόγω της μείωσης των καυσίμων και των ε, μορφών των καυσίμων που χρησιμοποιούνται. Αλλά αυτό έχει σχέση κυρίως με το πώς οργανώνονται τα σκάφη και φυσικά το διοξίδιο του θείου έχει επιπτώσεις ε, στο αναπνευστικό σύστημα, στα μάτια και ούτω καθεξής και αυτό το ποσοστό έχει σημαντικές συνέπειες για την υγεία μας. Για τον τομέα της ναυτιλίας τώρα, προσπαθούμε να δούμε και τι γίνεται και πώς ε, προχωρούν τα θέματα με τον ε, Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε και τι γίνεται. Ένα άλλο που μας ενδιαφέρει είναι η επιπτώση του θορύβου. Ο θόρυβος είναι ένας από τους πιο διεισδυτικούς έντονους παράγοντες στις πόλεις και στις αστικές περιοχές και 62% του πληθυσμού είναι εκτεσιμένοι στο μέσο όρο του θορύβου που είναι 55 δεσιμπέλ. Μέσο όρο. Τώρα, κατά τη διάρκεια της ημέρα, είναι σαφώς ένα πρόβλημα, διότι αυτό είναι ένα συγκριτικό στοιχείο που είναι ψηλό, ακόμα και αν το συγκρίνουμε με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εκεί που αυξάνονται τα στοιχεία, τα <clears throat> μετρήσαμε, είναι στην νυχτερινή έκθεση σε θόρυβο που έχουν αυξηθεί κατά 40% τα στατιστικά στοιχεία και έχουν σημαντικές επιπτώσεις ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Ο θόρυβος λοιπόν μας απασχολεί έντονα, μπορεί κανείς να ε, κατεβάσει από το διαδίκτυο ένα ε, ε, μέσο μέτρησης του θορύβου και να δείτε όλα αυτά τα, τα στοιχεία στο διαδίκτυο. Η επίτευξη των στόχων. Αυτή η έκθεση είναι η πρώτη αναφορά όσον αφορά ε, σχετικά με την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων ε, στην ναυτιλία λοιπόν ε, θέλουμε να επιτύχουμε 60% μείωση για, μέχρι το 2050. Ε, επίσης θέλουμε στα καύσιμα να έχουμε μία μείωση 40% μέχρι το 2050 και 95% μικρογραμμάρια μείωση των εκπομπών στα οχήματα. Τώρα, ε, αν σκεφτούμε τις μειώσεις στα καύσιμα μεταφορών, θα δούμε ότι υπάρχει 70% μείωση. Θέλουμε να επιτύχουμε μέχρι το 2050. 70%. Τώρα, για να προσεγγίσουμε αυτούς τους στόχους, αναλογιστήκαμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε, ποιο μπορεί να είναι το έναυσμα για να ξεκινήσουμε ε, σε έναν καλύτερο δρόμο. Βεβαίως ε, ε, ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε τις εναλλακτικές πηγές, υδροηλεκτρική ενέργεια, μεθάνιο, υγραέριο αλλά όλα αυτέ οι εναλλακτικέ ε, τα εναλλακτικά καύσιμα χρειάζονται υποδομή. Και η υποδομή πρέπει να εξασφαλιστεί. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν υπάρχει διείσδυση στην αγορά για τη δημιουργία αυτών των υποδομών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να χρησιμοποιήσουν τα εναλλακτικά καύσιμα. Ασφαλώς χρειαζόμαστε χρηματοδοτικά κίνητρα, ιδίω για την κατασκευή της, ε, των υποδομών. Και ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί ε, συνέχεια είναι η η επισήμαση, η επισήμαση η οποία αφορά ιδιαίτερα και ενδιαφέρει τους καταναλωτές. Θέλουμε την κατάλληλη επισήμαση ώστε να ξέρουν ότι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά καύσιμα, πιο καθαρά καύσιμα, καλύτερη ενέργεια, πιο αποδοτική και έτσι βελτιώνεται γενικά η κατάσταση. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα διαχωρίσει το, το θέμα της ανάπτυξης της οικονομίας και της ε, ανάπτυξης των μεταφορών. Δεν έχει γίνει ακόμα η αποσύνδεση αυτή, η οποία πρέπει να γίνει και ταχαίως. Γι' αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε σε μεγαλύτερη ζήτηση, σε οικονομική ανάπτυξη και σε, πιο, σε μεθόδους μεταφορών πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Άρα πρέπει σε όλους τους τομείς να αυξήσουμε την αποδοτικότητά μας. Οι μεταφορές ε, είναι ένας τομέας που δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Αυτό που λέμε στην έκθεση είναι ότι η αλλαγή των, μεταφορικών οδών και μέσων, η μετατροπή δεν σημαίνει μόνο μείωση των εκπομπών αερίων, αλλά σημαίνει ανταπόκριση και μείωση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι λαοί, οι πολίτες μας. Μπορείτε λοιπόν να δείτε αυτή την έκθεση. Αυτά είχα να σας πω εν περιλήψη και δίνω το λόγο σε εσά Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τα μέλη να μιλήσουν, να παρέμβουν. Η κυρία Αγιάλα Μάισεν και ο κ. Κράμερ. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Μαγκλέιτ για τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις σας και τα στοιχεία που μας δώσατε. Χαίρομαι που μας δίνετε πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Δύο ερωτήσεις πρώτον για το θέμα του θορύβου. Έχουμε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σύστημα αλλαγή ε, των ε, συστημάτων πέδωσης ε, για τα βαγόνια μεταφοράς εμπορευμάτων και εξετάσουμε κατά πόσον είναι αναγκαίο να ε, χρηματοδοτήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο στοιχίζει. Καταλαβαίνετε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχουν δυσκολίες αλλά μας το παρουσιάζουν ως το θαύμα των συστημάτων πέδησης. Δηλαδή, ε, πριν από αυτά τα φρένα και μετά από αυτά τα φρόνα, στις πόλεις τις οποίες περνούν τριάνα μεγάλους ε, έκτασης, ε, πλέον οι πολίτες θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι μετά από αυτή την εφαρμογή των συστημάτων. Θα μπορούσατε να μας δώσετε λοιπόν κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για το κατά πόσον θα υπάρξει σημαντική μείωση σε δεσιμπέλ και αν αυτή η μείωση είναι άνω ή κάτω των ποσοστών που μπορούν να αντέξουν οι πολίτες ε, στις διάφορες πόλεις. Ε, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τους ε, ε, ε σειρμούς τους οποίους ε, χρησιμοποιούνται. Και ένα άλλο ζήτημα είναι... αν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών αν γίνεται αλλαγή από αυτοκινητόδρομο σε τρένα. Διότι πολλές φορές ε, λέμε ότι ε, ε, είναι το θέμα του θορύβου, αλλά μας ενδιαφέρει και το θέμα της ρήπανσης ε, και υπάρχει σχέση και με την πηγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία λοιπόν για το τι γίνεται με τη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο, αν χρησιμοποιούνται περισσότερο σιδηρόδρομοι. Η κυρία Μάιστα. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ κύριε Μακλέιντ για την παρουσίασή σας τα ΔΕΔ τα, και οι κατευθυντές γραμμές, γραμμές τις οποίες θα συζητήσουμε μας δίνουν την ευκαιρία να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και να προωθήσουμε καλύτερα την επέκταση και τη διεύρυνση των σιδηροδρομικών μεταφορών, της ναυσιπλοείες κλπ. Είπατε πολύ σωστά ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον τομέα των μεταφορών. Ασφαλώς και στην εσωτερική αγορά χρειαζόμαστε απολύτως ε, ε τις Είπατε ότι ηλεκτρική, ε, τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα δεν έχουν αναπτυχθεί όπως τα θέλατε. Πράγματι, ακόμα και τα, η χρήση του υγραερίου ε, στα αυτοκίνητα δεν, είχε, δεν έχει τόσο ανέβει όσο θα θέλαμε. Είπατε ότι η ζήτηση είναι μικρή, μικρότερη της αναμενόμενης. Πέστε μας τις προοπτικές. Και δεύτερον, όσον αφορά τα σκάφη και το, ε, το υγρό καύσιμο, τα υγρά καύσιμα, είπατε ότι δεν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα καύσιμα τα πλοία και γι' αυτό ρηπαίνουν τόσο πολύ. Ορισμένα έχουν το ε, υγροποιημένο αέριο το οποίο το χρησιμοποιούν και ε, το παράπονο είναι, μάλλον ε, το εμπόδιο είναι η έλλειψη σταθμών ε, ε, λήψης του υγροποιημένου καυσίμου. Ναι, ναι, ναι. Η έλλειψη ενός δικτύου σταθμών εφοδιασμού. Υπάρχει προοπτική ανάπτυξη τέτοιων σταθμών. Ιδίω στην Βόρεια Θάλασσα που θέλουμε να μειώσουμε ε, ε, τη ρήπανση, συζητούμε την ε, εγκατάσταση πλυντηρίδων. Ο κύριος Κράμερ, ευχαριστώ τα, τα 30 δις τα οποία κερδίζουν οι ευρωπαϊκέ εταιρείε επειδή απαλλάσσονται από του δασμού τη κυροζήνη. Αναφέρεται πάρα πολύ ο ορισμό αυτό και δείχνει ότι η μέσο των μεταφορών από το 1990 έχει αυξηθεί 25% και βεβαίως έχει επιτευχθεί τεράστια πρόοδος. Οι συνθήκες ε, πλαισίου πρέπει να αλλάξουν. Τι μπορείτε να κάνετε από αυτού. Ε, εάν δεν αλλάξουμε ε, το πλαίσιο λειτουργίας, το το, το πλαίσιο ανάπτυξης δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, διότι συνεχώς επιβαρύνονται επιβαρυνόμαστε λόγω των μεταφορών. Είναι θέμα, μην ξεχνάτε, και ταχύτητος. Ε, Φοιτητέ οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν το τρένο βιάζονται και χρησιμοποιούν ε, τα αεροπλάνα, αερομεταφορές. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Γερμανία λέει όταν παρακολουθήσεις την αλυσίδα από την παραγωγή στη χρήση τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα υπολείπονται των προτύπων τα οποία είχαμε θέσει και μπορούμε ακόμα και κατά 25% να μειώσουμε την επιβάρυνση από τα αυτοκίνητα εάν βελτιώσουμε ε, τις ελλείψεις. Έχετε κοιτάξει όλη αυτή την αλυσίδα από την παραγωγή στη χρήση, στην κατανάλωση δηλαδή. Έχουμε επίσης διαπιστώσει στο Κοινοβούλιο ότι ε, πρέπει να αναφέρουμε ξεχωριστά για κάθε τρόπο μεταφορών τις, τα στοιχεία των εκπομπών. Μπορούμε, έχουμε διαπιστώσει, να μειώσουμε στην πηγή, ε, ιδίως στις συνδρομικές μεταφορές, ε, έχουμε το ένα κόστος μετατροπής 3,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό μας έχουν ε, τεθεί 10 ε, δισεκατομμύρια έχετε να μας ενημερώσετε ο εισηγητής κουνάει ήδη το, το κεφάλι του σίγουρα μπορούμε στην πηγή, στην κατασκευή να επιτύχουμε πολλά περισσότερα παρά συνεχίσει στις επόμενες φάσεις Επίσης το θέμα του θορύβου. Εάν ξυπνήσω τρεις φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας από ένα δυνατό θόρυβο, ε, εντάξει, μπορεί να, να επιζήσω. Όμως, τι γίνεται όταν έχω έναν συνεχή θόρυβο ε, όταν ας πούμε καίγεται, καίγονται τα πόδια μου και παγώνει το κεφάλι μου, μπορεί τα γόνατά μου να έχουν μια, ε, το μέσο όρο θερμοκρασίας. Μην κοιτάμε λοιπόν ε, με μονομένες μετρήσεις θορύβου, να κοιτάμε το μέσο όρο και τη, συνεχή καμπύλη. Και αυτό το οποίο θεωρώ σωστό είναι ότι αναφέρεται στις αερομεταφορές όχι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα αλλά και τις άλλες λιπογόνες ουσίες για τις οποίες οι ευρωπαϊκές εταιρείε είναι πολύ φιδωλές και δεν αναφέρουν πολλά στοιχεία. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε όλες τις μεταφορές πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο κίνησης, την κινητικότητα. Όπως είπατε, επαναλαμβάνω, οι μεταφορές δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Κινητικότητα, ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Κοπενχάγη τα τελευταία 20 χρόνια μειώθηκε σημαντικά η κίνηση των οχημάτων 300 αυτοκίνητα σε χίλιους κατοίκους. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι δυνατή η μετατόπιση προς άλλες, σε άλλους μεταφορικούς τρόπους, πέραν δηλαδή των αυτοκινήτων. Υπάρχει δυνατότητα. Ο κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε κυρία Αγγλέ για αυτή την παρουσίαση. Πιστεύω ότι το κίνητρο για τη μείωση των εκπομπών διευσυντήτου του άνθρακα είναι κατανοητό, απαραίτητο και ένα ευπρόσδεκτο εγχείρημα για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και πιστεύω ότι αντικατοπτρίζεται πολύ καλά στις τρέψεις εργασίες του Κοινοβουλίου αλλά δεδομένων στις πρόσφατες ε, απόφασης του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας να αναβαθμίσει την προειδοποίησή του για τις εκπομπές diesel ε, που ως πιθανού καρκινογόνου με παρόμοιες επιπτώσεις όπως το παθητικό κάπνισμα θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι το τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο για τον έλεγχο των εκπομπών κινητών οχημάτων και η ενθάρρυνση του πετρελαίου αντί για τις βενζίνες αντιμετωπίζει ουσιαστικά αυτά τα, ε, αυτούς τους ανησυχίες για την υγεία επαρκώς ή κατά πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι άλλο και αν ναι, τι. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος. Ε, περιμένετε λίγο. Η κυρία Γιάλα. Sí, justamente mientras... Ναι, ήθελα να επιμείνω λίγο. Αν μπορεί η κυρία Μαγκλέιτ να μας εμβαθύνει λίγο το θέμα της μείωσης των ε, ορίων ταχύτητας, διότι διάβασα στην έκθεσή σας ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν θετικά στοιχεία, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ε, ε, κάποια στοιχεία δεν είναι και τόσο θετικά. Θα μπορούσαμε λοιπόν στις συστάσεις που κάνουμε για τη μείωση των ορίων ταχύτητας να προσθέσουμε και το θέμα του θορύβου, διότι πολλές φορές οι κυβερνήσεις το χρησιμοποιούν για προεκλογικούς λόγους, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Να έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία, διότι φαίνεται ότι μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες για να έχουμε περισσότερα επιχειρήματα υπέρ τη μείωση των ορίων ταχύτητα. όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, αλλά και για λόγους υγείας. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Και εκ μέρου μου δύο παρατηρήσει κύριε ε, καθηγήτρια. Βρήκα πολύ ενδιαφερόντα τα διαγράμματά σα όσον αφορά τι εκπομπέ ε, τη ναυτιλία σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα. Ο Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός αποφάσισε να δημιουργήσει αυτές τις περιβαλλοντικές δράσεις για την ναυτιλία και δημιούργησε μία στη Βαλτική και μία στη Βόρεια Θάλασσα. Αλλά δεν δημιούργησε καμία τέτοια δράση για τη Μεσόγειο. Παρ' όλα αυτά Κοιτώντας τα εικόνες που μας παρουσιάσετε στις διαφάνειές σας, προκύπτει το ερώτημα για ποιο λόγο δημιούργησαν κάτι για τη Βαλτική και όχι για τη Μεσόγειο. Διότι εκεί έχουμε αυτή την κόκκινη περιοχή στο διάγραμμα. Εντάξει, και στη μάχη φυσικά υπάρχει πρόβλημα με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά εκεί φυσικά είναι αναμενόμενο διότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία πλοίων στη μάχη, αλλά αυτό που μας εκπλήσει είναι ότι επιλέγουν τη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα. Χωρίς να θέλω να πω ότι αυτό είναι λάθο, αλλά ουσιαστικά δεν πάνε εκεί όπου βρίσκεται το πρόβλημα σύμφωνα με τα διαγραμματά σας. Μπορείτε να μα σχολιάσετε. Το δεύτερο που ήθελα να πω αφορά την ρήπανση του αέρα. Με ενδιαφέρουν και οι τρεις πτυχές που αναφέρετε. Θέλω να σας προκαλέσω λίγο. Λέτε ότι η αεροπλοεία, η αεροπορία αντιπροσωπεύει το 4% και ότι στο σύνολό της ελάχιστα συνεισφέρει στις συνολικές εκπομπές. Ενώ το εκτιμώ αυτό και παρόλα αυτό, παρότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε τίποτα με την αεροπορία, Ουσιαστικά πού βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα ουσιαστικά είναι τα οχήματα επί των οδών, για να είμαστε ειλικρινείς. Όταν μιλάμε για τη Γλασκόβη, τη Γλασκόβη με τις υπερβολικές εκπομπές, έχουμε καθόλου νούμερα για το Λονδίνο, γιατί ακούω ότι το Λονδίνο πρόσκειται να ασκηθεί δίωξη στο Λονδίνο από την Επιτροπή επειδή δεν επιτυγχάνει τους στόχους ρήπανσης. Είναι σοβαρό το ζήτημα αυτό. Ε, ξέρω κατά πόσο συμφωνούν και ο κύριος Κράμερ και ο στη δική μου παρέμβαση, αλλά έχουμε λίγο χρόνο και θέλω να κάνουμε καλή συζήτηση εδώ. Μάικλ λοιπόν πρώτα και Φίλιπ. Κύριε Κράμερ. Ευχαριστώ. Βεβαίω, εδώ μιλάμε για αργό πετρέλαιο το οποίο χρησιμοποιείται στην ανοιχτή θάλασσα και θα πρέπει ουσιαστικά δηλαδή να εναποτίθεται ως, ως ειδικό απόβλητο, δηλαδή ειδικών ιδιωτήτων. Γιατί αυτό το καύσιμο, το αργό βαρύ πετρέλαιο δεν απαγορεύεται δεν απαγορεύεται. Ξέρουμε τι έρχεται επάνω μας, στις πλάτες μας, ε, γιατί δεν έχει ήδη τεθεί υπό απαγόρευση με τη χρήση άλλων ε, τι, ε, καυσίμων. Τι μπορείτε να μας πείτε από αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάω εξαιτία των όσων είπε ο κύριο Κράμερ, δύο σχόλιο. Μερικέ φορέ ακούγοντα τον κύριο Κράμερ, αναρωτιέμαι κατά πόσο θέλει να επιστρέψουμε στο να ε, οδηγάμε όλοι άλογα και κάρα. Α, αλλά τώρα δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι... Πολύ ωραία να το κάνετε λοιπόν αφού το θέλετε. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω. Το θέμα είναι κύριε Πρόεδρε ότι έχουμε δύο-τρία σημεία που ακούσαμε εδώ στη συζήτηση μέχρι στιγμή. Το ενδιαφέρον που ανέφερε ο κ. Κράμερ ε, ήταν η σύγκριση πόλεων όπως η Κοπενχάγη με τον ε, αριθμό, τεράστιο αριθμό ποδηλατών και σαν αναφέρεται και το Λονδίνο. Δεν συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Η Κοπενχαγή, για παράδειγμα, είναι πολύ μικρή πόλη σε σχέση με το Λονδίνο. Δεν μπορεί να αναμένει κανεί την ίδια κατανάλωση καυσίμων σε μια τεράστια μετρόπολη όπως το... σε μια τεράστια πρωτεύουσα όπως το Λονδίνο ή σε οποιαδήποτε άλλη πρωτεύουσα με 7, 8, 9 εκατομμύρια πληθυσμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε φορά που ακούω σε μια από αυτές τις συζητήσεις φαίνεται ότι η συζήτηση πολλώνεται μεταξύ δύο άκρων. Κάτε με, τέθηκαν δύο ζητήματα στην παρουσίαση και στη συζήτηση που ακολούθησε. Το πρώτο είναι η διαχείριση της ζήτησης. Κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια συζήτηση μιλάμε για διαχείριση της ζήτησης. Θα σας το πω καθαρά, εγώ δεν είμαι υπέρ της διαχείρισης της ζήτησης για να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη σε μια κατάσταση όπως τη σημερινή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να γνωρίζουμε, όπως είπε η κυρία Μάισνερ, ότι χρειαζόμαστε μεταφορές και χρειαζόμαστε τα αγαθά να φτάνουν στις αγορές. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα για μένα. Για μένα δηλαδή το ζήτημα είναι πώς με αποδεκτό τρόπο για το γενικό πληθυσμό μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα αγαθά θα φτάνουν στις αγορές. Το άλλο ζήτημα το οποίο αναφέρεται συχνά εδώ είναι η δαιμονοποίηση ουσιαστικά των οδικών μεταφορών. Στην πραγματικότητα οι οδικές μεταφορές για το προβλέψιμο μέλλον θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να μεταφέρουμε τα αγαθά στις αγορές. Μπορούμε να μιλάμε για μεταφορά για μετατροπή από οδικέ μεταφορέ στι σιδηροδρομικέ και όλα αυτά δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα για μερικά χρόνια θα χρειαζόμαστε οδικέ μεταφορέ, ειδικότερα σε περιοχές ε, ε, νησιωτικές που δεν ανήκουν στη ε, κύρια ε, Ήπειρο. Το επιχείρημα μου εδώ είναι ότι ναι, φυσικά θέλουμε να ασχοληθούμε με τις εκπομπές ρήπων. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και την πραγματικότητα και να δούμε τι είναι πραγματικά δυνατό και όχι τι είναι απίθανο. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας. Κύριε Γκλέιντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ασχοληθώ με το τελευταίο σχόλιο, διότι θεωρώ ότι αφορά και πολλές άλλες γενικότερε ερωτήσει που ακούσαμε στη συζήτηση. Αυτό που λέει αυτή η έκθεση είναι ότι τα συνεχή μοτίβα μεταφορών είναι τέτοια που δεν θα επιτύχουμε τους στόχους. Αν τα αντιμετωπίσουμε τμηματικά αυτά τα μοτίβα, δεν μιλάμε απαραίτητα για διαχείριση της ζήτησης. Αλλά λέμε περίπου ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μια κατάσταση μεγαλύτερων οδικών ταξιδιών για τους ίδιους σκοπούς, όπως σήμερα, δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό στο μέλλον. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό. Δεν είναι έλεγχος της ζήτησης, διότι εν τέλει, όταν μιλάμε για εμπορευματικές οδικές μεταφορές, βλέπουμε κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις ε, ουσιαστικά σύμπτυξης ε, αγαθών και οχημάτων και ε, μεταφορές πολλών αγαθών ταυτόχρονα και εκεί βλέπουμε αλλαγές. Αυτό λέμε ότι πρέπει να επισημανθεί ως σωστή πρακτική. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε για τις πόλεις. Φυσικά θα πρέπει να συγκρίνουμε παρόμοια πράγματα, αλλά αν κοιτάξουμε το Βερολίνο για παράδειγμα, κοιτάξτε την εκθέση της σελίδα 43 αργότερα, θα δείτε ότι όπου έχουν υλοποιηθεί περιοχές ε, μειωμένων εκπομπών επιτυγχάνονται μειώσεις που επιζητούμε. Δηλαδή είναι θέμα απόδοσης ε, και είναι και μια εικόνα του τι μπορεί να παρέχουν οι οδικές μεταφορές. Τώρα όσον αφορά την ταχύτητα, ξέρουμε ότι η επιβελή του νόμου τελικά αποτελεί τα στοιχεία κλειδιά με τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται, υλοποιούνται μεταφορές. Ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι οι εκπομπέ αερίων θερμοκηπίων πρέπει να είναι ένα από του στόχου που θα πρέπει να διατηρούμε στο στόχαστρο. Τώρα, όσον αφορά το χάρτη για την αυτιλία, δεν θέλω να υπάρχει σύγχυση. Στη Βαλτική μιλάμε για διοξίδιο του θείου. Στη Μεσόγειο μιλάμε για σωματίδια. Πρέπει δηλαδή να δούμε το χάρτη ω έχει στη Βαλτική ουσιαστικά ελέγχουμε το διοξίδιο του θείου για να καταλάβετε τώρα γιατί μιλάμε. Και αυτό είναι το ζήτημα. Το ίδιο ισχύει για την αεροπορία. Ναι, φαίνεται να είναι μικρές οι συνεισφορές ε, όσον αφορά το ε, ε, οξύδιο του αζότου, αλλά αν δούμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, φυσικά η αεροπορία είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να εστιαστούμε. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι σε θέματα ζήτησης ουσιαστικά ο τρόπος ανακατανομής των αγαθών σε ολόκληρη την Ευρώπη δημιουργεί πολλά προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά τις υδάτινες οδούς ε, και τη χρήση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς και αλλαγής τρόπων μεταφοράς, γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν προβλήματα για τη διατήρηση ορισμένων επιπέδων υδάτων στις θάλασσες μας και αυτό ουσιαστικά ε, αναφέρει ότι τα επίπεδα των υδάτων μπορεί να μην είναι τα ίδια με το παρελθόν. Τίποτα λοιπόν δεν είναι δεδομένο όταν μιλάμε για αξιοποίηση πόρων και υποδομών. Και απλά θέλω να το θέσω αυτό ως δεδομένο. Θα ήθελα να ζητήσω από τον συναδελφό μου να απαντήσει δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Την πρόταση για το θόρυβο και τα συστήματα πέδησης. Τον ειδοποιώ δηλαδή για το τι πρέπει να απαντήσει και για τις γραμμές για το TNT. Δεν είμαι σίγουρη για τις απαντήσεις για αυτό το θέμα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να πω ότι στη συζήτηση που είχαμε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι απολύτως σαφές ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποτελείται αυτή τη στιγμή από συντηρητικές κατά κάποιο τρόπο επιτροπές θεωρώντας ότι το ντιζέλ είναι καρκινογόνο. Η νομοθεσία μας είναι επαρκής. Όχι, δεν είναι. Και είναι πρόκληση για εμάς τώρα αυτό Αφενός περιμένουμε μία ε, αρχή αξιόπιστη να έχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να προχωρήσει αυτή την κατηγοριοποίηση αλλά χρειάζεται αρκετός καιρός γι' αυτό και είναι απολύτως σαφές ότι είναι η έκθεση σε όζων και όλους τις πρόδρομες ουσίες που σημαίνει ότι υπάρχει έκθεση του πληθυσμού σε επίπεδα πολύ ανώτερα από τα ωραία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Τώρα στην έκθεση για την ποιότητα του αέρα μπορείτε να τα δείτε αυτά λεπτομερώ. Μπορείτε να δείτε τι εκθέσει δηλαδή των αστικών πληθυσμών σε όλα αυτά. Θα ήθελα τώρα να σα ρωτήσω, Αλφρέντο, αν μπορείτε να μα μιλήσετε γρήγορα για τα συστήματα πέδηση και κατά πόσο έχουμε ε, ε, scrubbers στην Βαλτική και όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Για τα θέματα του θορύβου, υπήρξαν κάποιες νέες εξελίξεις στην νομοθεσία, η οποία θα συζητηθεί τώρα. Υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο τομέα στον οποίο θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι. Πρόκειται για ε, σταδιακές βελτιώσεις, οι οποίες λίγο-λίγο θεωρούμε ότι θα βελτιώσουν τα επίπεδα του θορύβου στις πόλεις. Δεν έχω διαβάσει την πρόταση για τα συστήματα ε, πέδησης ε, που μειώνουν ουσιαστικά το θόρυβο των σύρμων στους σιδηροδρόμους, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν εξελίξεις σε αυτό. Όσον αφορά τώρα τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, Υπάρχουν κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Ένα από τα σημαντικά είναι η φραγμή στη συνεργασία μεταξύ χωρών για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων. που έχουν συνέπεια. Όταν έχουμε υποδομές για διάφορες μορφές μεταφορών, είναι σίγουρα κάτι το οποίο μπορεί να έχει ε, μείωση και στη ρήπανση και στα αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου η αλλαγή από τις οδικές αρτηρίες σε άλλα μέσα μεταφοράς σίγουρα έχει θετικές συνέπειες και φαντάζομαι ότι στις κατευθυντήριες γραμμές ε, οι προτάσεις που έχουμε θα οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να τις εξετάσουμε λίγο πιο επισταμένα. Το Δεκέμβριο θα γίνει και η παρουσίαση του πράσινου διαδρόμου στο Μάλμο. Ε, αυτό θα είναι ένα από τα σημεία τα οποία μπορούμε να εξετάσουμε αν έχουμε εφαρμογή αυτών στην πράξη. Και θα αξιολογήσουμε και όλο το πρόγραμμα για να δούμε πού έχουμε προστιθόμενο όφελος ε, σε σχέση με την αλλαγή που γίνεται. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου. Ευχαριστώ. Ναι, κάτι ακόμα, η κυρία Μακλέιτ. Να δούμε αν μπορούμε να έχουμε μια πλήρη αλυσίδα, μια αλλαγή στα ε, αυτοκίνητα οχήματα. Υπάρχουν πολλά προϊόντα στην αγορά Ακούσαμε και επιχαίους τίτλους από μη κυβερνητικέ οργανώσεις για το τι χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένα αυτοκίνητο, αλλά στην, ε, στον κόσμο των υλικών αρχίζουμε να έχουμε μια μεγάλη αλλαγή, όχι μόνο σε θέματα ανακύκλωση, διότι μα ενδιαφέρει ο κύκλο ζωή ενό οχήματο ε, και τα ανταλλακτικά του, αλλά υπάρχουν τάσει ε, για πιο ελαφρά αυτοκίνητα με καλύτερα υλικά και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να δω λοιπόν κατά πόσον το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να δεχτεί την ιδέα να κάνουμε μία μελέτη για το πώς ακριβώς ε, είναι ένας κύκλος ζωής παραγωγής ενός αυτοκινήτου οχήματος ε, και κατά πόσον χρησιμοποιούνται και ενετόμες τεχνολογίες. Ε, εάν το Κοινοβούλιο λοιπόν ενδιαφέρεται να το εξετάσει λίγο πιο σοβαρά, εμείς μπορούμε κάλλιστα να βοηθήσουμε με τους συναδέλφους από το Κοινό Κέντρο Έρευνας που ασχολούνται με τα θέματα αυτά μια ερώτηση εκτός μικροφώνου. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό αυτή τη στιγμή, απαντάει η ομιλήτρια. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να τεθεί, αλλά δεν έχουμε απάντηση προς το παρόν. Δυστυχώ δεν μου απαντήσατε. Τρεις ρώτησα. Ε, πώς θα εξελιχθεί η αγορά αυτοκινήτων, ηλεκτρική ενέργεια, ε, υγραέριο, όσον αφορά τι πλυντηρίδε, και τις εγκαταστάσεις ίσως είναι πολύ τεχνολογικό και λεπτομερές το θέμα, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό μπορεί να συνδεθεί με το θέμα των ε, εκπομπών ε, διότι υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ε, διάφορα ορυκτά για την πλήση, για τη λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων. Και λυπάμαι που δεν μου απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Θα μπορούσατε να επανέλθετε σε αυτά. Ναι, φυσικά κύριε Πρόεδρε, ήθελα να επανέλθουμε για τις πλυντρίδε, γιατί δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση τώρα όσον αφορά τα διάφορα καύσιμα και τις διαφορέ επιπτώσει που είπατε για το Ρότερνταμ, όπου θέλετε να χρησιμοποιούμε πλοία μηδέν εκπομπών. Υπενθυμίζουμε τώρα ότι με τη Γενική Διευθύνση ΜΑΡΕ εξετάζουμε την καλύτερη δυνατή ε, διαδικασία ώστε να περάσουμε σε καθαρές εκπομπές, καθαρό στόλο, ώστε να υπάρχουν ευκαιρίες όχι μόνο για τα ίδια τα σκάφη, αλλά και στον τρόπο διαχείρισης του ίδιου του πλοίου και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να το επισημάνουμε αυτό κατά τις εργασίες μας μέσα στο επόμενο έτος και να επανέλθουμε σε εσά μια καλύτερη εικόνα του θαλάσσιου στόλου. Είναι κάτι το οποίο θα είναι το αποτέλεσμα τη παρουσία Τώρα, όσον αφορά τα ύδατα, πρέπει να σα πω: Κάνατε πολλέ ερωτήσει, για τι οποίε δεν έχουμε συγκεκριμένε απαντήσει. Τι έγραψα όλε εδώ και σίγουρα θα επανέλθω σε εσά με κάποιε απαντήσει. Ευχαριστώ. Okay. Ευχαριστώ. Εφόσον, εάν μπορείτε να απαντήσετε γραπτός, εντάξει. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Μαγκλέιντ και τους συναδέλφους της ε, για την παρουσίαση της έκθεσης και την ανταλλαγή απόψεων και προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία. Πέντε λεπτά, πέντε λεπτά να αλλάξω την καρέκλα μου που έχει σπάσει και με πονάει τη μέση. Okay, colleagues, can we now, it's 10 o'clock, can we now move on to... Ο Πρόεδρος, μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα για να, στην ψηφοφορία να κάνουμε τώρα έναν έλεγχο της τεχνολογίας καταρχάς. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία για τον έλεγχο των καρτών και του συστήματος. Wait for Mr. Ertug to sort out his many credit cards from his voting card. Περιμένουμε να ξεχωρίσει ο κύριος Σίτοκ τι ε, τις του κάρτες από την, την κάρτα ψηφοφορίας του. Ωραία. Ψηφίσατε πέρα τη ψηφοφορία Για να δούμε. δεν έχει ξεπεραστεί, δεν μας περισσεύει καμία ψήφος, είναι όλες εντάξει στον αριθμό, λοιπόν, συγχαρητήρια. Okay. We'll start with the draft report on... Αρχίζουμε με το σχέδιο έκθεσης για την πρόταση μιας οδηγίας, τροποποίηση οδηγίας 16 του 2009 για τον έλεγχο του κράτους λιμένος.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 Ήταν γλωσσική λοιπόν τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται η 32. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συγγνώμη, η 33 απορρίφθηκε και η 34. 2 υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τη 2 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, ήταν σαφή σαφέστατο, αλλά για λόγους ευγένειας, όχι. Ναι, απορρίφθηκε, απορρίφθηκε, εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Όταν η γραμματεία μου λέει ότι είναι σαφές το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έξι αφορά μόνο την παράγραφο 5 του άρθρου 18 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 καταπίπτει. 9 υπέρ ε, έχει μια τεχνολογική φύσεως. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 καταπίπτει α όχι το 10 είναι ακόμα πρέπει να ψηφιστεί υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά, άποχες, δεκτή. 16 υπέρ. Το 40 καταπίπτει γιατί έγινε δεκτή 15. 16 υπέρ. Κατά άποχες. Δεκτή. 17 υπέρ. Κατά άποχες. Δεκτή. 41 υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 44 προφορική τροπολογία από τους συντάκτες. Υπάρχει αντίρρηση στην προφορική τροπολογία όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 44 με την ε, προφορική τροπολογία. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Η 45 έχει αποσύρθει. 46, 47, 48 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. ψοφήσατε όλοι, πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτονται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 20 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος 22 ε, άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 24 την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροποποιηθήσα πρόταση. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 35 υπέρ, 4 κατά. Και την, το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίζουμε τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Το ψήφισμα, το ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε η ψηφοφορία. Το ίδιο ακριβώ. 35 υπέρ, 4 κατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης ε, στην πρόταση για οδηγία που αφορά τις ευθύνες κράτους σημαίας και την εφαρμογή της ε, ε, οδηγίας 13 του 2009. Προτείνουμε να τα ψηφίσουμε όλα μαζικά. Έχει κάποιος αντίρρηση γι' αυτό. Δεν το δέχονται. Ας δούμε λοιπόν μια με τροπολογίες. Οι δύο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία τέσσερα υπέρ, σαράντα συγγνώμη, κατά, αποχές, εγκρίνεται. σαράντα ένα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. έξι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για 9 με ψηφοφορία κατά τμήματα που ζήτησε το άλλο το πρώτο κομμάτι και το δεύτερο uncertification. Πρώτο κομμάτι λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 με 16 μπορούμε να ψηφίσουμε μαζικά. Όχι, εντάξει. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά,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 Ψήφισαν άπαντες, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρινέται με 34 υπέρ, καμία κατά, 5 αποχές συγχαρητήρια. Κύριε Μπαχ. next. Ακολουθεί η ψηφοφορία για το ε, κανονισμό ΕΜΣΑ, μία ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 34 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Φλέγκενστάιν. Ωραία, έτσι ολοκληρώνεται αυτό το κομμάτι της συνάντησης. Περνάμε τώρα στη συνεδρία των συντονιστών.